αφορά την αίτηση των Ολλανδικών αρχών για την άσκηση της ασυλίας του κ. Κράτσμαν βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6 παράγραφος 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραπευθεί αυτή η αίτηση στην νομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δεύτερη